προσφύγων στις προαναφερθήσεις χώρες. Προχωρούμε στην ψηφοφορία. Πρόκειται για την απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση προσωρινών μέτρων στα πλαίσια της διεθνούς προστασίας υπέρ Ιταλίας, Ελλάδος και Ουγγαρίας. Έχω λάβει ορισμένες τροπολογίες από την ομάδα EFDD. έχει, έχει υποβάλει ορισμένε απορριπτικέ τροπολογίες και θα δείτε ότι έχει και ορισμένες υπέρ των οποίων τις οποίες είναι θετικές. υπέρ. Ερχόμαστε πρώτα στο άρθρο 2α. Ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορίας. Απερίφθη. Η τροπολογία υπαριθμών 6 με ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία υπαριθμών 7 με ονομαστική ψηφοφορία επίσης αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι και όλες. Πέρας. Απορρίπτεται και αυτή. 8 δέλτα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Πέρας. Απερίφθη. 9 δέλτα. Με ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απερίφθη. 10 δέλτα, πάλι ονομαστικά, αρχίζει. Ψηφίζατε όλοι. Πέρας. Απερίφθη. 11 δέλτα. Ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει. Ψηφίσατε. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 4, πάλι ονομαστικά. Ψηφίσατε. Πέρας. Απερίφθη. Ερχόμαστε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει η ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε ψηφίσατε Ψηφίσατε 556, 370 υπέρ, 134 κατά και 52 αποχές. Σχέδιο νομοθετικού περιεχομένου ψηφίσματος. Εδώ έχω την τροπολογία υπαριθμών 3. Κοινή τροπολογία πλειών πολιτικών ομάδων. Ψήφι παρακαλώ υπέρ με το χέρι. Ανατάσχυρος. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σύμφωνα με το σχόλιο 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. το νομοθετικό περιεχόμενο ψήφισμα ονομαστικά, παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Κυρίες και κύριοι, τα πρακτικά